Έχω να σας δώσω διά, διάφορες ε, πληροφορίες. Καταρχάς, σας παρακαλώ να καθίσετε όλοι, ούτως ώστε να ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας. Γιατί έχουμε πολλά σημεία στη μερίσια διάταξη. Έχουμε ήδη καθυστερήσει, μάλιστα. Να σταματήσουν τα πηγαδάκια, παρακαλώ. Κάποιες πληροφορίες που θα ήθελα να σας δώσω λοιπόν. Την επόμενη εβδομάδα, την ε, Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου, από τις 6 ε, μέχρι τις 7, μπορείτε να συμμετάσχετε στην τρίτη συνεδρίαση, τη διαθεσμική για τις πληρωμές. Θα είναι πάρα πολύ σημαντική, μια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μία ενημέρωση για τις πληρωμές ε, για το Πουδουπού 2014-2020 καθώς και για την περίοδο μετά το 2020. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνεδρίαση λοιπόν. Στις 18 Οκτωβρίου λοιπόν. Ζητώ συγγνώμη αλλά κάνετε πάρα πολύ θόρυβο. Παρακαλώ καθίστε. Ας προσπαθήσουμε να ησυχάσουμε. Στις 18 Οκτωβρίου θα γίνει και ένας ε, τρίλογος στην, για τα δημοσιονομικά και η διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υποστηρίξει τις ε, τροπολογίες που έχουν υπο, ε, υιοθετηθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών πριν δύο εβδομάδες. Να υπενθυμίσω ότι η Ολομέλεια θα ψηφίσει τη θέση της για τον προπολογισμό του 2018 στην επόμενη Ολομέλεια στις 25 Οκτωβρίου. Μετά από αυτό θα ξεκινήσει η περίοδος ε, συνδιαλλαγής και κάποια από τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών θα υποδειχθούν από την πολιτική του ομάδα για να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής. Αυτό, αυτοί πρέπει να σημειώσουν ότι η πρώτη σύνοδος της Επιτροπής Συνδιαλλαγής θα γίνει τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου στις 3.30 ε, ώρα και η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής θα συνεδριάσει από τις 2.30 ώρα για να προετοιμάσει αυτή τη θέση. Επίση, σημειώστε ότι η δεύτερη σύνοδος της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, δεύτερη συνεδρίαση, συνεδρίαση που μπορεί να κλείσει ενδεχομένως τι διαπραγματεύσεις, θα γίνει στις Βρυξέλλες την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου. Στο τέλος της ε, εβδομάδα τη Ολομέλειας ε, του Νοεμβρίου του Στρασβούργου. Και εάν δυστυχώς, αν τελικά δεν οδηγηθούμε σε αποτέλεσμα, θα φτάσουμε μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, τόσο ώστε να κλείσουμε έτσι αυτή την ε, συνδιαλλαγή. Επίσης, οι συντονιστές συνεδρίασαν χθες, θα ήθελα να σας πω, ούτω ώστε να ευθυγραμμιστούμε με τις ε, υποχρεώσεις ε, διαφάνειας που δεσμεύουν και τις άλλες επιτροπές και οι συζητήσεις των συντονιστών θα οδηγούν σε ένα προσάρτημα το οποίο θα προσαρτάται στις, ε, στο... στη μέση διάταξη. Και μόνο οι επίγουσες αποφάσεις ε, θα σας ε, διαμηνύονται στην αρχή της συνεδρίασης. Οι αποφάσεις για τους χθεσινούς διορισμούς είναι ότι η ομάδα της ΚΟΕ έχει αποσύρει το αίτησή του. Οι συντονιστές λοιπόν αποφάσισαν ότι ο πρόεδρός σας θα αναλάβει την προετοιμασία της νομοδότησής μας για την Επιτροπή ΑΦΕΤ για το, την εφαρμογή των εξωτερικών μηχανισμών πληρωμής ε, ενδιάμεση αναθεώρηση μέχρι το 2020 και, την, ε, και τις μελλοντικές πληρωμές μετά το 2020. Επίσης θα ασχοληθώ με την γνωμοδοτή για την ΕΚΟΝ, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, για τις οικονομικές πολιτικές, ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών. Επίσης οι συντονιστές αποφάσισαν ότι ε, θα ετοιμάσουμε την γνωμοδότηση της ΜΠΑΤΣ για τις ε, υπηρεσίες τραπεζικής εποπτείας, για τους ε, φορείς μάλλον τραπεζικής εποπτείας. Επίσης, λάβατε μία ανακοίνωση για τα πρακτικά, του σχεδίου πρακτικών, της συνεδρίασης της 29ης Ιουνίου. Έχετε παρατηρήσεις και αν όχι, θεωρώ ότι εγκρίνονται. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, Γιάς Γκάιερ. Έχουμε ένα σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 6 για τον προπολογισμό 2017. Η Κομισιόν ετοίμασε, παρουσίασε χθε ένα σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού για να προσαρμόσει ε, τα έσοδα του προπολογισμού, όπω γίνεται κάθε φορά τέτοια εποχή, ε, στα πλαίσια τη εκτέλεση του προπολογισμού, με βάση τι εκτιμήσει ε, που κάνουμε για του διάφορου ίδιου πόρου. Μία αναθεώρηση προ τα πάνω των ποσών που εισέπαξε η Κομισιόν 2,2 δισεκατομμύρια. Και κάτι άλλο που συμβαίνει για δεύτερη συναπτή χρονιά, να μειώσουμε τις πιστώσεις πιστώσεων, πληρωμών μάλλον, λόγω του ότι έχουμε υποπληρωμές στην πολιτική συνοχής. Μιλάμε ε, για ένα συνολικό ποσό 7,7 ε, δισεκατομμύρια ευρώ για, το, για τις πιστώσεις ε, της πολιτικής συνοχών. η Κομισιόν παρουσίασε πριν από λίγες μέρες ένα ποσό για τις μη χρησιμοποιηθήσεις πιστώσεις που έχουν φτάσει σε ένα σημαντικό επίπεδο. Μιλάμε για 682 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Ιουρέλ, ο οποίος είναι διευθυντής, θα μπορούσε να μας πει δύο λόγια για αυτό το ποσό. Για το συνολικό ποσό, καθώς και για τα 682 εκατομμύρια. Ευχαριστώ. Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού που προτείνει η Κομισιόν έχει τρία στοιχεία. Όπως είπε συνοπτικά ο Πρόεδρος, το πρώτο στοιχείο είναι μια πολύ σημαντική μείωση των ε, πληρωμών που προτείνεται ε, σε ένα συνολικό ποσό 7,7 δισεκατομμύρια. Αυτό κατανέμεται ε, σε διάφορους τομείς, όχι στον 1α όμως, που θα τον ενισχύσουμε στις συνολικές μεταφορές πιστώσεων, αλλά όλοι οι υπόλοιποι τομείς θα πρέπει να υποστούν μείωση του, των πιστώσεων πληρωμών. Όπως είπε ο Πρόεδρος, η πιο σημαντική μείωδος ε, είναι στο 1β για την πολιτική συνοχή, δηλαδή η Κομισιόν προτείνει μία μείωση 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι σε απόλυτη ευθεία γραμμή με την ε, ε, μείωση των προβλέψεων των κρατών μελών που έχει λάβει η Κομισιόν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τέλος Ιουλίου και αυτή η μείωση που υπέδειξαν τα κράτη-μέλη τα ίδια συμπεριλαμβάνει και μια μείωση 5,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επομένως λοιπόν υπάρχει απόλυτη ευθυγράμμιση με αυτό που μας είπαν τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία για το χαμηλό επίπεδο εφαρμογής και εκτέλεσης και ο Επίτροπος Έτιγκερ θα κάνει ε, μία παρέμβαση στην επόμενη, την επόμενη εβδομάδα και στον τριμερή διάλογο και στη διαθεσμική συνάντηση για το θέμα των πληρωμών. Και θα είναι τότε μια ευκαιρία για να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Η δεύτερη μείωση αφορά το τομέα 2. Το θέμα της ανάπτυξης. Δεν είναι και τόσο επίμαχο αυτό το θέμα. Αυτές είναι πληρωμές που καταφέραμε να κάνουμε στο τέλος του 2016 μετά την μεταφορά πιστώσεων που γίνεται στο τέλος της χρονιάς. Ε, αρχικά αυτές οι πληρωμές ε, θα γινόταν το 2017, αλλά έγιναν τελικά προκαταβαλικά ε, το 2016. Μιλάμε για 0,8 δισεκατομμύρια που μπορούμε να απελευθερώσουμε υπό το τομέα 2. Επίσης, στον τομέα 3 υπάρχει μείωση. Την ανακοίνωση Κομισιόν πριν το καλοκαίρι είπε ότι θα υπάρχει μια υποεφαρμογή, υποεκτέλεση, Έχουμε χρησιμοποιήσει τμήμα αυτού του πλεονάσματο για να χρηματοδοτήσουμε την, τις πληρωμές στο DAB5, στο Διορθωτικό Προπολογισμό 5, ε, για το EFSD. Επίσης, έχουμε χρησιμοποιήσει το πλεόνασμα για να χρηματοδοτήσουμε την ε, μεταφορά 18 για το ITER. Ο κύριος Γκάιερ το σχέδιο γνωμοδότησής του για τον Διορθωτικό Προπολογισμό 5 αν κάνει συγκεκριμένη μνήμα στο θέμα αυτό. Επομένως, υπάρχει μια μικρή υποεφαρμογή την οποία προτείνουμε να ξαναδώσουμε πίσω. Τέλος, για τον ε, τομέα 4 προτείνουμε να επιστρέψουμε 0,7 δισεκατομμύρια από τα προενταξιακά εργαλεία και από το μηχανισμό γειτονίας για διάφορους λόγους. Φερρυπίν, ε, ε, το μηχανισμό για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, παρότι ο μηχανισμός αυτός προχωράει καλά, οι πληρωμές όμως έχουν καθυστερήσει λόγω περίπλοκων διαπραγματεύσεων για τις, μεγάλα έργα υποδομών. Σε ό,τι αφορά το μηχανισμό για τη γειτονία, υπήρχε ένα πρόβλημα καθυστερήσεων ε, προς διάφορες χώρες, ε, Αίγυπτος, Μαρόκο, Μολδοβία, Αρμενία και Ατζερμπαϊτζάν. Γιατί τα κριτήρια εκταμίευσης δεν έχουν τηρηθεί. Και αυτό προκαλεί καθυστερήσεις. Τέλος, η Κομισιόν προτείνει να επιστρέψει, να δώσει τις πιστώσεις που αφορούν την προχρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν έχουμε λάβει καθόλου αιτήσει για προχρηματοδότηση και επομένως όλα αυτά τα λεφτά μπορούν τώρα να απελευθερωθούν. Το δεύτερο στοιχείο του σχεδίου προϋπολογισμού αφορά την προσαρμογή των ιδίων πόρων και τις πληρωμές αυτές που κάνουν τα κράτη-μέλη στον προϋπολογισμό, ε, συνολικά υπάρχει ουδετερότητα, δεν επηρεάζει δηλαδή το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού και τα ποσά, αλλά έχουμε μεταφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη ποσών, πιστώσεων δηλαδή, ε, ώστε το τελικό αποτέλεσμα είναι μηδέν, ουδέτερο. Η Κομισιόν προτείνει τα, οι πληρωμές των κρατών μελών να ευθυγραμμιστούν με τις πιο προ... τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις. Αυτό είναι μία άσκηση που γίνεται κάθε χρόνο. Επίσης, υπάρχει μια πρόταση για αναθεώρηση του υπολογισμού της ε, μείωσης ή επιστροφής ε, του, για, το Ευρω... για το Ηνωμένο Βασίλειο ε, για τα έτη 2016. Το τελικό στοιχείο του διορθωτικού προπολογισμού είναι αύξηση του ποσού των προστήμων. Από σήμερα η Κομισιόν έχει λάβει το τελικό ποσό των προστήμων, 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ και μια και στον προϋπολογισμό είχαμε προβλέψει μόνο 1,1 δισεκατομμύρια, Μπορούμε να προσθέσουμε 2,1 δισεκατομμύρια στη χρηματοδότηση του προπολογισμού, που αυτό μειώνει επίση την ανάγκη να συνεισφέρουν ποσά τα κράτη-μέλη. Η συνολική επίπτωση λοιπόν του διορθωτικού προπολογισμού για τι συνεισφορέ των κρατών μελών θα είναι από τη μία μία μείωση των ε, πιστώσεων πληρωμών κατά 7,7 δισεκατομμύρια και από την άλλη μία μείωση λόγω τη ε, αύξηση ε, του ποσού των προστήμων πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Συνολικά τα κράτη-μέλη θα χρειαστεί να πληρώσουν λιγότερα 9,8 δισεκατομμύρια στους ίδιους πόρους. Για το συνολικό ποσό που μεταφέρεται, μιλάμε για 680 εκατομμύρια που θα μεταφερθεί με, μεταξύ διαφόρων ε, δημοσιονομικών γραμμών για την ενίσχυση όμως πάντα του τομέα 1α. Προτείνουμε λοιπόν διάφορες μειώσεις σε άλλους τομείς ε, που χρεια... για πολλές γραμμές του προϋπολογισμού όλες θα πάνε για να τροφοδοτήσουν τον τομέα 1α. Αυτή η ενίσχυση γίνεται για να ενισχύσουμε την, το, ε, της, ε, το Ταμείο Εγγύησεων, το Χειρικό Ταμείο Εγγύησεων. Να τροφοδοτήσουμε λοιπόν αυτό το Ταμείο με 150 εκατομμύρια. Επίσης, περισσότερες πληρωμές χρειαζόμαστε για τα διάφορα ε, προγράμματα ε, παροπλισμού των πυρηνικών σταθμών. Χρειαζόμαστε μια ενίσχυση των πληρωμών για ασφαλείς μεταφορές και για τον Γαλιλαίο. Υπάρχουν διάφορες μειώσεις επίσης που μπορέσαμε να εντοπίσουμε ότι χρειάζονται. Οι πιο σημαντικές είναι η αλία, τομέας 2, γιατί και εδώ υπάρχει πρόβλημα κοινοποίησεων της ε, υπόδειξης των αρμοδίων αρχών δεν έχουν υποδειχθεί ποιε είναι οι αρμόδιε αρχέ γενικά στην Αλία. Ε, τομέα 4 έχουμε κάποιε μειώσει που μπορούν να γίνουν στο εργαλείο αναπτυξιακή ε, συνεργασία και στα πλαίσια τη μακροοικονομική βοήθεια και κάποιε μειώσει εντό του 1α που αφορούν τον ορίζοντα 2020, το κόσμο Ελπίζω να σας δώσω μια σφαιρική αλλά λακωνική εικόνα ε, για τις προτάσεις αυτές. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ. Κύριε Γκάιερ, θέλετε να πάρετε το λόγο να μας πείτε τις δικές σας εκτιμήσεις. Ευχαριστώ και σύντομα κύριε Πρόεδρε. Διότι ήδη εδώ και 15 λεπτά θα έπρεπε να έχει αρχίσει η ψηφοφορία κανονικά. Κυρίε και κύριοι, αυτή η υπολοιπόμενη ε, εφαρμογή ή υποεφαρμογή αν θέλετε ε, είναι ανισχυτική. Έχουμε μια δυστυχώς γνωστή κατάσταση. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση την οποία γνωρίζουμε που αξίζει να συζητηθεί και να αναλυθεί περισσότερο που θα κάνω όμως, θα ξεκινήσω τη συζήτηση αυτή με τον εισηγητή Ζίκφριντ είτε τα ζητούμενα ποσά από τις χώρες μέλη είναι υπερβολικά υψηλά από την αρχή και δεν μπορούν να απορροφηθούν από τις χώρες γιατί έχουμε μετά ένα και έχουμε μάλλον μετά ένα πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις ή υπάρχει κάπου αλλού ξεφεύγει από κάπου αλλού η διαπραγμάτευση. Τέλος πάντων είναι διαφορετικές οι προτεραιότητες που πρέπει να συζητηθούν και επανεξεταστούν. Συνήθως η διαδικασία που ακολουθεί η παρούσα Επιτροπή είναι να τίνει να βάζει περισσότερα χρήματα σε μια γραμμή του προπολογισμού για μια πολιτική προτεραιότητα από ό,τι θεωρούν ίσως σωστό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες μέλη για να δείξουμε ότι είναι δικός μας πολιτικός στόχος. Αλλά τα χρήματα αυτά μετά δεν απορροφώνται. Και αυτό ενδεχομένω οφείλεται σε διοικητικέ αδυναμίε των χωρών μελών. Αυτό με ανισχύει ακόμη περισσότερο βέβαια, διότι εκεί μπορεί να έχουμε τελικώ ένα πρόβλημα σε σχέση με το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Γίνεται λοιπόν όλο και μεγαλύτερη η αδυναμία αυτή, όσο περισσότερο οι χώρε μέλη δεν είναι σε δυνατότητα να δαπανίσουν τα χρήματα αυτά. Και είναι ένα στρατηγικού χαρακτήρα το πρόβλημα αυτό, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή. Θα, πρέπει εξάλλου να εξεταστεί, όταν δηλαδή βλέπω τι προτάσει που γίνονται στην κατηγορία 2, για την ανάκτηση χρημάτων. Αν αυτά έχουν σχέση περισσότερο με το γεγονός ότι οι διοικήσεις των χωρών μελών δεν οργανώνουν σωστά την διαχείριση των χρημάτων, ή αν οφείλεται περισσότερο στο ότι μειώνεται η ζήτηση χρημάτων για τους πρόσφυγες. Αυτό είναι κρίσιμο για το τι θα γίνει παραπέρα με την συγκεκριμένη γραμμή του προϋπολισμού. Προετών δεν προλαβαίναμε να ικανοποιήσουμε τις ε, απαιτήσει των χωρών μελών για τα θέματα αυτά. Και τώρα είναι η δεύτερη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αφαιρεθούν χρήματα από την κατηγορία 3, από AMF και ε, SMF και να, μπουν, να σε άλλες κατηγορίες. Ε, εδώ πρέπει να εξετάσουμε πρώτα ποιες είναι οι αιτίες και μετά να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα. Θα το κάνω εγώ αυτό στην έκθεσή μου, σε συνεργασία με τους ε, συναδέλφους μου. Θα πω κάπως αόριστα μεν, αλλά θα καταλάβει ο συγκριτή εννοώ ότι θα πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση αυτή σε σχέση και με τις διαπραγματεύσεις με τους μελλοντικού προπολογισμού. Δεν θέλω να πω τίποτε τώρα καταληκτικά, γιατί θα τα κάνουμε αυτά μέσα στην προπαρασκευή του επόμενου τριμηρού διαλόγου. Σε ό,τι αφορά τώρα το DAB6, τον, ε, το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού, υπάρχει μεταφορά πιστώσεων, με έχει ενημερώσει η γραμματεία ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος για να συζητηθεί περαιτέρω η, το σχέδιο εκθέσεώς μου. Αυτό είναι κάπως ατυχές, αλλά θα βρούμε πιστεύω κάποιο άλλο τρόπο και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε συμφωνία. Όμως κάπου κάπου θα πρέπει να διαθέτουμε χρόνο για να μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση σε περισσότερο βάθος. Ευχαριστώ πάντως κύριε Πρόεδρε. Θέλει κάποιος το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να θέλει κανείς το λόγο. Ο κύριος Μούρεσαν, Γενικός Εισηγητής για το 2018. Εν συντομία, κύριε Πρόεδρε, χωρίς να καταχραστώ πολύ του χρόνου, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες, αυτό το σχέδιο τροποποίησης του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει ότι η θέση μας για τον προϋπολογισμό της Ένωσης για την επόμενη οικονομική χρήση είναι η σωστή. Στο 1α θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα, να προχωρήσουν τα έργα, η ζήτηση είναι υψηλή, πρέπει να το ενισχύσουμε το 1α και να μην περικοπεί κατά 750 εκατομμύρια ευρώ όπως προτείνει το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού το δικό του. Τώρα, ως προς την υποεκτέλεση του προϋπολογισμού πρέπει να σκεφτούμε κύριε Πρόεδρε ποια είναι η καλύτερη μορφή να λύσουμε το ζήτημα, να το αντιμετωπίσουμε συστηματικά. Η υποεκτέλεση θα οδηγήσει σε προβλήματα στα τέλη του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Οι συσκέψεις για τις πληρωμές αρκούν σαν μορφή, σαν σχημά. Ή μήπω πρέπει να το αναθεωρήσουμε μετά από τις αντιδράσεις των κρατών μελών στα σχόλια της Επιτροπής. Νομίζω ότι πρέπει να λειτουργήσουμε πιο συστηματικά, να βρούμε πιο συστηματικό και πιο εντατικό τρόπο ορισμένα κράτη-μέλη τα πάνε καλά, αλλά άσχημα να δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς μπορούμε να συστηματικοποιήσουμε αυτή την προσέγγιση, να έχουμε ενδεχομένω ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για να βελτιωθούν οι προβλέψει. Αυτά κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ενδιαφέρον θα ήταν να έχουμε ένα κατάλογο αναχώρα για να δούμε ποιες χώρες δυσκολεύονται περισσότερο από τις άλλες. Ακούω στη χώρα όπου εκλέγουμε για παράδειγμα ότι ε, πολλοί παρετούνται από, το, από κονδύλια του Ταμείου Συνοχής γιατί τα προγράμματα είναι τόσο περίπλοκα και διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς προτιμούν να παρετηθούν από αυτά από το να υποχρεούνται να ε, συμπληρώνουν φακέλους εξαιρετικής περιπλοκότητας για να ε, τύχουν χρηματοδότησης. Άρα να τα διαφωτίσουμε όλα αυτά και η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να αναθέσει τη τις μελέτης της επόμενης εβδομάδας, ακριβώς για να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει, συμβαίνει με αυτή την υποκατανάλωση των ε, κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής για να αντιληφθούν και τα κατάλληλα διδάγματα για το επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αν δεν θέλει κάποιο άλλο το λόγο, θέλω να σας πω ότι ο Γενικός Εισηγητής θα μας παρουσιάσει, ο κ. Γκάιερ, το σχέδιο της έκθεσής του για το έκτο διορθωτικό σχέδιο του προεπολισμού την επόμενη εβδομάδα και ότι το γενικότερο έμβασμα των 6, τόσο ε, εκατομμυρίων ευρώ θα αποτελέσει αντικείμενο ψηφοφορία στην Επιτροπή μας σε λίγα λεπτά. Και γι' αυτό τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη ψηφοφορία, να μπούμε στην ε, φάση των ψηφοφοριών. Θα ήθελα να βάλετε τις ηλεκτρονικές κάρτες στο μηχάνημα για να κάνουμε μια ε, δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε. Ψήφισαν όλοι. Λείπουν τρεις ψήφοι. Τρεις που δεν ψήφισαν. Ένας, μία ψήφος λείπει. Κάποιος έχει βάλει την κάρτα του αλλά δεν έχει ψηφίσει. Όχι, όχι, δεν μιλώ για τον εαυτό μου. Ξέρω ότι ε, πλεονάζω, περισσεύω. Η δική μου ομάδα είναι υπερβολικά παρούσα, όπως πάντοτε. Καλώς, 35. Πριν ψηφίσουμε λοιπόν το σχέδιο ψηφίσματος για το σχέδιο τροποποίησης του προϋπολογισμού για το 2018, όπως ε, συντάχθηκε από τον κύριο Μουρέσα να σας δώσω το λόγο στον Γενικό Συγητή, τον κύριο Μούρεσαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να πω. Το ψήφισμα αντικατοπτρίζει πλήρως αυτά που ψηφίσαμε πριν από δύο εβδομάδες για τη θέση του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό και τις σχετικές τροπολογίες χρειάστηκε να περιορίσω το ψήφισμα σε αυτό και να περιορίσω το, τον όγκο των πολιτικών σχόλειων και ε, σχολιασμών που δεν σχετίζονται με το 2018. Η προτεραιότητά μας ήταν σαφής καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, η αντίδραση στη θέση του Κοινοβουλίου επίσης, άρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο να προσθέσω προς το παρόν. Ευχαριστώ. Ακούγονται κλάματα μωρού, δεν φαντάζομαι. Όντω είναι λίγο βασανιστικά αυτά που λέμε. Το παραδέχομαι. Παρακαλώ, συνεχίστε. Το κατάλαβα το μήνυμα κύριε Πρόεδρε, το πιασα. Και γι' αυτό ολοκληρώνω κάπου εδώ, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ. Καλώς. Ψηφίζουμε λοιπόν για το σχέδιο ε, του ε, ψηφίσματος. Λοιπόν, συμβιβαστική υπαριθμών 1. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Υπερψηφίζεται η συμβιβαστική 1. Τροπολογία 6. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18 αποσύρεται. 19. Πρώτο τμήμα του 19. Ψηφίζουμε. Το δεύτερο καταπίπτει. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το πρώτο μέρος το 19. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 αποσύρεται. 22 υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για το 27. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Όχι, αποσύρεται 31. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 56 τροπολογία. Καταπίπτει. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62. Καταπίπτει. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 και 80 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά. Αποχές θα επαληθεύσουμε για της ηλεκτρονικής οδού. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 82 παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 23-15. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Το δεύτερο τμήμα της 97 ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λείπει μία ψήφος. Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 19 υπέρ 18 κατά και μία αποχή. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 101. Τροπολογία 101 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 102. Τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχ... Όχι, κατά πίπτη ζητώ, ζητώ συγγνώμη. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Άποχες νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά πρέπει να το ελέγξουμε. Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 111. Πέρας. Απορρίπτεται, όντως, 23-15. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Όχι, καταπίπτει. Συμβιβαστική 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 125 καταπίπτει. 126 επίσης. 127 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 128 και 129 ίδιο αντικείμενο υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ Κα, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 136 και 137 με ίδιο αντικείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 136 και 137. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτονται. 138 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. 139 και 140 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 141 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το, η 142 καταπίπτει, 143 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται η τροπολογία. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 145. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Σας παρακαλώ να σηκώνετε το χέρι. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 153. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 155-156 δύο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έχουμε μία προφορική τροπολογία του εισηγητή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για τα άλλα τμήματα τώρα από την τροπολογία 160 ή 160 καταπίπτει, 161 ψηφίζουμε προφορική τροπολογία του εισηγητή ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 164 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 165 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται νομίζω, αλλά θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινούμε ηλεκτρονική ψηφοφορία την 166. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100... Συγγνώμη. Την 167 θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Καλώς. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 167. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 168 κατά πίπτη. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 173. 173 το λόγο έχει ο συγητής, παρακαλώ. Όχι εσείς. Ο κύριος Άσουορθ. Ναι. Είναι μια προφορική τροπολογία, Πρόεδρε, αλλά την έχετε πάρει και έχετε την εξήγηση μπροστά σας. Είναι μια τροπολογία που έχει να κάνει με λεπτομέρειες και στοιχεία που μας δίνει η Γενική Διεύθυνση Finance και τις λεπτομέρειες τις έχετε στη γραπτή επεξήγηση που σας έχει μοιραστεί. Ψηφίζουμε λοιπόν την 173 την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά. Δεν είναι σαφές ποιος είναι υπέρ της 173 με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται αλλά θα το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. δεν ήταν καθόλου προφανές. Γιατί τα χέρια σας δεν τα σηκώνατε. Εγκρίνεται. 174 υπέρ. Κατά. Ποιος είναι κατά του 174, της 174. Αποχές. Απορρίπτεται 175 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 177 καταπίπτει 178, 179, 180, 181 καταπίπτουν επίσης 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 183 κατά πίπτη. 184 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται, 185 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται, 186 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται, την 186. Η 187 καταπίπτει. Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 186. Ζητώ συγγνώμη. Ξεκινάμε και την ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Την 186. Ψηφίσατε όλοι. Ε, εγκρίνεται. 187 καταπίπτει. 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 189 υπέρ κατά δεν είναι σαφές ψηφίζουμε την 189 ηλεκτρονικά πέρας απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία. 190 πήδη 191 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 192 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Πάμε στις νομοδοτήσεις των διαφόρων επιτροπών. Άφετ 9 υπέρ Κατά. εποχές, Υιοθετείτε. Ίντα. Κοντ. Πάμε στην κοντ 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Έκον ε, 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Έκον 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Θα ζητήσουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση για την κοντ 15. Ψηφίστε τώρα. Πέρα ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. 21 ψήφι υπέρ, 17 κατά. MB13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Ήτρε. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Ρέτζι. 8. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείται άγκρι 18 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται πες 5 θέλετε παλήθευση της άγκρι 18 ψηφίστε τώρα ΠΕΣ ψηφοφορίας υιοθετείται 20 υπέρ, 14 κατά. Πες 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Καλτ 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Καλτ 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τελειώσαμε τελική ψηφοφορία, με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 30 ψήφι πέρ 6 ψήφι κατά και 2 εποχές. Ευχαριστώ τον γενικό εισηγητή και τον ειδικό εισηγητή, τον κύριο Ashworth. Και τώρα πάμε σε ένα ψήφισμα για το έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ψήφισμα που ετοίμασε ο κύριος Ολμπριχτ και η κυρία Τουμά. Τροπολογία 3, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβασμός α υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 23, τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές θα το επαληθεύσουμε αυτό το σημείο ηλεκτρονικά. Πέρας προφορίας για την τροπολογία 23. 18-18. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24. αποσύρεται. 25 αποσύρεται. Συμβαστική B. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Θα την επαληθεύσουμε αυτή ηλεκτρονικά. Την 37. Πέρας φοφορίες. Απορρίπτεται. 20 ψηφί κατά, 13 υπέρ, 39 υπέρ. Κατά. Άποχες. Νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά επειδή σηκώνει το χέρι, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για επαλήθευση. Ψηφίζουμε την 39. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφόριας. Απορρίπτεται. 20 κατά 12 υπέρ. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41. Με μία προφορική τροπολογία. Και ψηφίζουμε σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά, αποχές. Υιοθετεί το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. υιοθετείτε Τροπολογία 42, υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 43 και 44, ίδιος στόχος, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 48 υπέρ κατά αποχές θα την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 48 ψηφίσατε όλοι όχι λείπει μια ψήφος πέρας προφορίας Υιοθετείτε. 21 ψήφι υπέρ, 15 κατά, 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική C υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική D υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 57 αποσύρεται. Συμβαστική Ή. E, υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Τροπολογία 67 καταπίπτει. Η 68 επίσης καταπίπτει. Πάμε στην 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 72 υπέρ κατά θα επαληθεύσουμε την 72 ηλεκτρονικά ψηφίσουμε τώρα ψηφίσατε όλοι πέρας προφορίας απορρίπτεται 21 ψήφικα κατά 15 υπέρ. Συμβαστική F. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Συμβαστική G. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Υιοθετείτε. Συμβαστική H. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβαστική I. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Υιοθετείτε. Τροπολογία 1. Αποσύρεται. Η 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για το σύνολο του κειμένου ψηφίζουμε τώρα με ηλεκτρονική ψήφο. Ψηφίζουμε τώρα. Παρακαλώ. Πέρας προφορίας. Εγκρίνεται. 20, 27 ψήφοι υπέρ, 6 κατά. Συγχαρητήρια στους δύο συγκητές. Κύριε Γκέιερ, μας παρουσιάσετε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού του 2017 για τη χρηματοδότηση το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Μπορούμε να ψηφίσουμε on block. Μπορούμε. Εάν δεν έχετε αντίρρηση. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε. Για να εξοικονομήσουμε και λίγο σάλιο. Κατά. Αποχές. Αυτές οι τροπολογίες καταρρύπτονται. Ε, καταπίπτουν. Ψηφίζουμε συνολικά το κείμενο ηλεκτρονικά τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας προφορίας. Εγκρίνεται. 31 ψήφοι υπέρ, 4 κατά και 2 εποχές. Τώρα, για την κινητοποίηση του Μηχανισμού Ευελιξίας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμη ανάπτυξη. Μία ηλεκτρονική ψήφος, δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ξεκινάει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 31 ε, ψήφι υπέρ, 5 ψήφι κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στην Πιογκάγη. Έκθεση για την εφαρμογή της πολιτικής ΚΕΠΑ. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά θα την επαληθεύσουμε την 5 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε τώρα. Ψήφισατε όλοι. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Πέρας φοφορίας. Υιοθετείτε 20, 21 ψήφι πέρα 14 κατά. Τροπολογία 6 πέρ Κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ψηφίσουμε τώρα πέρας προφορίας απορρίπτεται 18 ψήφοι κατά, 17 υπέρ. Η 7 ήταν αυτή, έτσι δεν είναι. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Για το σύνολο του κειμένου με η χρονική ψηφοφορία. Ψηφίσουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας προφορίας. Εγκρίνεται. 25 ψήφι υπέρ, 10 κατά, μία αποχή. Πάμε τώρα στο συνολικό ποσό που αναφέρθηκε. από τον κύριο Ιουρέλ, τον Διευθυντή της, Γενικής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Διευθύνσης Badge της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν θέλει ο Γενικός Εισηγητής, θα ψηφίσουμε το ποσό αυτό για την πρώτη πληρωμή. Πληρω... Ε, ψηφίστε τώρα με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Πέρας προφορίας. Εγκρίνεται 26 ψήφοι υπέρ, 4 κατά και 2 εποχές. Τώρα ψηφίζουμε. Το ΤΕΚ 25 ε, βοήθεια για την Ιεμένη. Ο κύριος Σιουρέλ θα μπορούσε να μας ε, πει δύο λόγια για αυτή την πληρωμή. Και μετά ο γενικό Συγητής, ο κύριος Γκάιερ, θα πάρει το λόγο. Κύριε Ιουρέλ, δύο λόγια παρακαλώ για το ΔΕΚ 25 και 26. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γκάιερ, τον Γενικό Εισηγητή για την αποδοχή της πρότασης αυτής. Δέχτηκε να το ψηφίσουμε πολύ γρήγορα το σημείο αυτό, γιατί η Κομισιόν έστειλε την πρόταση ή τις προτάσεις πριν λίγες μέρες μόλις στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ τον εισηγητή λοιπόν που κινήθηκε τόσο γρήγορα γιατί αυτές οι δύο προτάσεις είναι κατεπίγουσες. Τα μέλη της Επιτροπής βλέπουν ότι προσπαθούν να ανταποκριθούν σε δύο ανθρωπιστικές κρίσεις και ιδίω στην Ιεμένη και την Αιθιοπία. Για την Ιεμένη και στις δύο περιπτώσεις η Κομισιόν προτείνει ε, την κινητοποίηση της μεταφοράς του αποθεματικού κατεπίγουσας βοήθειας προς το ανθρωπιστικό μηχανισμό γιατί η εφαρμογή του ανθρωπιστικού μηχανισμού από τα τέλη Σεπτεμβρίου είναι 96% σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις ε, υποχρεώσεων και έχουμε μόνο 50 εκατομμύρια στο αποθεματικό για αυτό το εργαλείο. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτήσουμε τις ε, κατεπήγους ανθρωπιστικές δράσεις από τις συνήθεις πιστώσεις. Γι' αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε από το αποθεματικό για την κατεπήγουσα βοήθεια. Για την Ιεμένη προτείνουμε 25 εκατομμύρια σε υποχρεώσεις επιπλέον των 52 εκατομμυρίων που είχαν, είχαν δοθεί νωρίτερα το 2017 μέσω του προπολογισμού της Ένωσης για να χρηματοδοτήσουμε ε, βοήθεια που σώζει ζωές και την χρειάζεται η χώρα, ε, τρόφιμα, γιατί υπάρχει χολέρα αυτή τη στιγμή στην Ιεμένη και για να χρηματοδοτήσουμε επιμελητιακή υποστήριξη για την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας για την Αιθιοπία. Η Κομισιόν προτείνει ένα ποσό 15 εκατομμυρίων σε υποχρεώσεις ε, που αφορούν κυρίως ε, την κατάσταση της διατροφικής ανασφάλειας που επιδεινώνεται γοργά και θα μπορούσε να φτάσει σε ακραία επίπεδα στην Αιθιοπία εάν δεν δοθεί επιπλέον βοήθεια υπάρχει μια παρατεταμένη ξηρασία που οδήγησε σε σημαντική απώλεια ζώων. Περίπου 2 εκατομμύρια ζώα χάσαμε και αυτό μείωσε την πρόσβαση των οικοκυριών στα τρόφιμα. Επιπλέον η κατάσταση ε, επιδεινώνεται λόγω φοβερής επιδημίας ε, χολέρας. Ευχαριστώ τον εισηγητή λοιπόν που δέχτηκε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύο επίγουσες ε, του επίγοντε αυτούς φακέλους πολύ γρήγορα και ελπίζω και η Επιτροπή, τα μέλη δηλαδή με την ψηφοφορία τους, με την ψήφα τους να δεχτούν αυτές τις δύο προτάσεις. Ευχαριστώ τον εισηγητή, ο κ. Γκάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ιστορικό εξηγήθηκε. Εν ώψη των πολύ απειλητικών αυτών θεομηνιών, κρίσεων, καταστροφών, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και είναι αναγκαίο να υπερψηφιστούν ταχύτατα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Άρα, η ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει. Τέλος. 28 ψηφιπέρ, 2 κατά και 1 αποχή. Το λόγο λαμβάνει ο κύριος Τάραντ για τρει μεταφορές πιστώσεων για άλλα τμήματα του προϋπολογισμού 2017. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα δύο πρώτα, οι δύο πρώτες δηλαδή είναι εύκολες. Αφενός για την διευκόλυνση δραστηριοτήτων των βιβλιοθηκών με νέες τεχνολογίες, 4 και 5, και να ψηφίσετε υπέρ. Η τρίτη ωστόσο είναι προβληματικότερη, διότι όχι για πρώτη φορά φέτος, το συγκεκριμένο θεσμικό όργανο ζητεί περισσότερα χρήματα για επικοινωνίες. Και με αυτές τις επικοινωνίες εννοεί μάλλον να χρηματοδοτεί τα μίντια να τα να δωροδοκεί τα μίδια και να οργανώνει ευχάριστες συναντήσεις. Θέλω λοιπόν να σας ζητήσω μία εβδομάδα παραπάνω για να εξετάσω καλύτερα το θέμα και σας ζητώ αναβολή της πληροφορίας για σήμερα. Ευχαριστώ. Καλά λοιπόν, για τις δύο πρώτες μεταφορές εκφραστήκατε θετικά δεν είναι αναγκαίο να ψηφιστούν. Μπορώ να θεωρήσω λοιπόν ότι εγκρίνονται. Και νομίζω ότι αφού δεν υπάρχει και επίγον χαρακτήρας όπως εξηγήσατε και εσείς κύριε Σιγητά, μπορούμε να συμφωνήσουμε μαζί σας και να αναβάλουμε την ψηφοφορία για το ΔΕΚ 1 2017. Και επανέρχομαι στην πολιτική ακινήτων. θέμα όπου προβλέπεται να προσθεθούν δύο εβδομάδες στην αξιολόγηση για την πολιτική κινήτων. Η κυρία Χόλμα έχει συναντηθεί με τους κοιόδης ηγητές και με τους υπεύθυνου των ε, οργανισμών. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Κύριε Πρόεδρε, Οι σκιώδες και εγώ ασχοληθήκαμε εντατικά με το θέμα της μίσθωσης ακινήτου στο Λουξεμβούργο. Και θεωρούμε, θεωρούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην διαδικασία. Ως εισηγήτρια, αλλά και οι συναδελφοί μου, θεωρούμε ότι μας θέτουν πρώτα τελεσμένο γεγονότα ή μάλλον μας ασκούν πιέσεις που δεν μπορούμε να δεχτούμε και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί. Θα σημειώσω επίσης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι, αγαπητοί κύριε Διευθυντά, δεν είναι παραδεκτή από μας τέτοια στάση εκ μέρους σας και αναμένω από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών να έχει πρώτα-πρώτα στη διάθεση του προσωπικού κατάλληλα, κατάλληλους χώρους γραφείων και όχι της δεκαετίας του 70 και τρίτο να τα κάνει αυτά με τρόπο που να ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες ανάγκες. Τα λέω αυτά σύντομα και διπλωματικά διότι πραγματικά έχω θυμώσει πολύ με τον φάκελο αυτό. Καλούμαστε να λάβουμε απόφαση για τους συνεργάτες της Επιτροπής στο Λουξεμβούργο για τα κτίρια δηλαδή που αναγκάστηκαν πράγματι να εγκαταλείψουν ε, με πολύ σύντομες προθεσμίες διότι ανακαλύφθηκε αμίαντος ε, στα κτίρια αυτά. Είπαμε βεβαίως η υγεία υπερτερεί απέναντι οποιοδήποτε κόστους, αλλά ακόμα αναζητούν τα κατάλληλα κτίρια. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Πράγματι, διαρθρωτικά και παρακαλώ την πρόεδρο τώρα της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού, κυρία Γκρέσλε, να παρακολουθήσει τη λέω, διότι η δομή έτσι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί. Μιλούμε για χώρους αποθηκών που μας κοστίζει το μίσθωμα σε βάση χρόνου 500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον οι ελάχιστες προϋποθέσεις ασφάλειας, διότι πάνε να χώσουν τους ανθρώπους αυτούς να εργαστούν σε κτίρια που δεν υπάρχουν καν έξοδοι κινδύνου για περίπτωση πυρκαγιάς. Πραγματικά μπαίνουν σε κίνδυνο οι ζωές των ε, συνεργατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω πραγματικά αγανακτήσει. Αντιλαμβάνομαι βεβαίω τις ανάγκες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν καταλαβαίνω όμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν έρχεται και λέει ότι οφείλει να μισθώσει ακίνητα στο Λουξεμβούργο. Πρώτο θα πρέπει να εξεταστεί η δομή εάν πραγματικά χρειάζεται να αποθηκεύει προϊόντα όπως καφέ, ρύζι και άλλα σε αποθηκευτικούς χώρους. Δεύτερο, όταν έχουμε εκτυπωτήρια. Οι συνεργάτες και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων που είναι κατεστημένα στο Λουξεμβούργο, όπως το δικαστήριο κλπ. Να χρησιμοποιούν τα ίδια τους ίδιους εκτυπωτές αυτά είναι παροχές υπηρεσιών και δεν επιτρέπουν στους μεν να χρησιμοποιήσουν τις εκτυπωτές των δε. Πολύ ευχαρίστως δηλαδή φαίνεται πως κάνουν επικάλυψη δύο και τρεις φορές. Διότι φαίνεται πως δεν τους απασχολεί καθόλου το κόστος. Ζητώ λοιπόν και από την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και γι' αυτό παρακαλώ τα λόγια μου να σημειωθούν στα πρακτικά, να εξεταστούν οι διαθρώσεις αυτές στο Λουξεμβούργο. Ασφαλώς και χρειάζεται να μισθωθούν, να μισθωθούν κτίρια στο Λουξεμβούργο. Αν όμως δεν βρίσκουν τους κατάλληλους χώρους και αν το κράτος του Λουξεμβούργου δεν είναι διατεθειμένο να βρει αποθηκευτικούς χώρους, θα έλεγα τότε να φύγουμε από το Λουξεμβούργο. Αν δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει χώρος. Και σας λέω και καθαρά, τα κτίρια στο Βέλγιο κοστίζουν τρει φορέ λιγότερο. Κοστίζουν το 1 τρίτο του μισθώματο από αυτά που καλούμεθα να πληρώσουμε στο Λουξεμβούργο. Βρίσκω δηλαδή ολόκληρη αυτή τη διαδικασία πραγματικά ένα σκάνδαλο. Αν θέλει το Λουξεμβούργο να εκπληρεί την, ε, ε, τα προπροπόμενα συνθήκη, δηλαδή να εγκαθίσταται ένα μέρο του προσωπικού των κοινοτήτων εκεί, θα πρέπει να προσφέρει του κατάλληλου χώρου. Εάν όχι, δεν είμαι διατεθειμένη στο μέλλον να εγκρίνω ούτε μία δεκάρα δαπάνες. Θα πω λοιπόν να φύγουμε από εκεί. Για αποθευτικιστικό χώρο με 500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα για ένα χρόνο. Ακόμα και το κανονικό μίστομα για ε, κτίρια κατοικίας δηλαδή είναι 280, 280 ε, ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και 180 εδώ στις Βρυξέλλες, στο κέντρο των Βρυξελών. Εν τέλει πραγματικά σας ομολογώ δεν ήξερα καν τι να κάνω και με εκπλήσει το γεγονός ότι και το Συμβούλιο Υπουργών το οποίο έρχεται και μας κάνει προβλήματα και για την τελευταία δεκάρα, το τελευταίο λεπτό του ευρώ, δεν θέτει καν ερωτήσεις για το θέμα. Δεν αντιλαμβάνομαι τι κάνουν οι υπηρεσίες του Συμβουλίου όταν καλούνται να ελέγξουν το θέμα. Παρακαλώ λοιπόν τους συναδέλφους μου να κατανοήσουν αυτή τη δυσαρέσκεια την οποία νομίζω εκφράζω αρκετά καθαρά. Βέβαια δεν βλέπω και άλλο τρόπο παρά να εγκρίνουμε για την πενταετία αυτή. Αλλά λέω καθαρά στην Κομισιόν. Σε πέντε χρόνια θα πρέπει να έχει ξεκαθαριστεί η αλλαγή των δομών. Θα πρέπει να είναι καθαρό ποια θεσμικά όργανα εγκαθίσταται στο Λουξεμβούργο και γιατί. το να διατηρούμε εκεί κάποιε υπηρεσίε μόνο και μόνο επειδή έχουμε την συμβατική υποχρέωση απέναντι στο Λουξεμβούργο δεν το αντιλαμβάνομαι. Και στα πλαίσια τη γνωμοδότηση έχω σημειώσει με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο τα όσα λέω. Δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα στην πενταετία. Αυτό όμω που επικρίνω εντονότατα είναι ότι τον Ιούνιο μα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το κτίριο, το μελλοντικό κτίριο Ζαμονέ είναι απολύτω εντάξει. Στο μεταξύ μαθαίνω εντελώ συμπτωματικά 1,5 χρόνο μετά, ότι χρειάζονται νέα μέτρα για την ασφάλεια. Έστω το δέχομαι, αλλά να μας τα πούν τότε από την αρχή, διότι εμείς λάβαμε απόφαση το 2013, στην οποία απόφαση λέει ότι το κτίριο Ντρόσμπαχ, όπου πάμε τώρα να νοικιάσουμε, να μισθώσουμε νέα τμήματα, είχαμε ζητήσει με την απόφασή μας να εγκαταλειφθεί το κτίριο αυτό διότι το μίστομα είναι υπερβολικά υψηλό. Τώρα πάνε να νοικιάσουν και άλλα τμήματα του Ντρόσπαχ επειδή λέει δεν βρίσκουν αλλού. Να με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, έπρεπε να τα πω αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή, διότι ομολογώ ειλικρινά ότι έτσι δεν είναι δυνατό να συνεχίσουμε. Δεν ενημερωνόμαστε επαρκώ ω Επιτροπή Προπολογισμών. Ε, ξαναλέω, τυχαία τα έμαθα τα πράγματα αυτά. Και παρακαλώ την DG Badge τη Επιτροπής να επεξεργαστεί τα θέματα αυτά πάρα πολύ προσεκτικά και πάρα πολύ γρήγορα. Να υποβάλει τις σχετικές εκθέσεις όσο γίνεται συντομότερα. Ευχαριστώ. Εγώ παρατηρώ ότι αυτός ο φάκελος και αυτή η υπόθεση έθεσε σε κίνδυνο την υγεία του εισηγητή. Δεν μου έχει ξανατύχει τέτοιο πράγμα, λέει η κυρία Χόλμαρη. Πρόκειται για πράγματα τριτοκοσμικά για, για χώρους όπου λέει αποθηκεύουν το ρύζι. Son expression orale était de nature à, à la libérer. Πράγματι, το γεγονό ότι είχατε την ευκαιρία να εκφραστείτε πιστεύω ότι σα ε, έκανε να εκτονωθείτε και να εκφραστείτε πραγματικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να φύγει ένα βάρο από πάνω σα. Η κυρία Καρθία Θαμπάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μπω στην ουσία του θέματος, γιατί η πολιτική για τα κτίρια και ειδικά η πολιτική για τα κτίρια στο Λουξεμβούργο θα έφτανε μόνη της για να φτιάξουμε σενάριο για μια σαπουνόπερα που θα κρατούσε χρόνια ολόκληρα. Σαπουνόπερα λέτε. Καλή διαχείριση. Εμείς αποφασίσαμε να επενδύσουμε εκεί που οι τιμές είναι πιο εφικτές, αλλά ίσως και οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί. Ίσως αυτό πρέπει να κάνουμε στο Λουξεμβούργο. Σε κάθε περίπτωση, λέει οι βουλευτές, θέλω να ε, σχολιάσω ένα θέμα διαδικαστικό επί της ουσίας. Χθες στις 7 το απόγευμα πήραμε αυτό το ψήφισμα και πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα. Ξέρω ότι είναι μια κούρσα, ένας αγώνας δρόμου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Ε, χθες Ευτέρα το βράδυ και να προλάβουμε να διαμορφώσουμε σωστή άποψη και είναι ένα επίσημο παράπονο και θέλω να το διατυπώσω. Ο Πρόεδρος, καταλαβαίνω την παρατήρησή σας, όμως πριν από δύο εβδομάδες ήδη ασχοληθήκαμε με αυτή την υπόθεση. Ναι, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα. Θα πρέπει να έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε. Δηλαδή το διαβάσαμε εντάχει σήμερα το πρωί όσο συζητούσαμε για άλλα στην Επιτροπή. Το διαβάσατε. Ναι. Κοιτάξτε έγινε μια κοινή συνεδρίαση με τους σκιώδεις εισηγητές που δεν μπόρεσαν να συμπαριστούν και τους διαφόρους συνεργάτες και είπαμε τα βασικά. Δηλαδή, περιγράψαμε την κατάσταση, ασκήσαμε κριτική, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε άλλη επιλογή πρέπει να πάρουμε μια θετική απόφαση. Στη συνέχεια ήμουν άρρωστη για μια ολόκληρη εβδομάδα, άρα από την Παρασκευή Ήμουν καθυλωμένη στο κρεβάτι και έπρεπε αυτά να τα συντονίζω από το ε, κρεβάτι, γιατί ήμουν άρρωστη. Εστάλησαν όλες οι πληροφορίες τους και οι εισηγητές. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστερημένη αποστολή ε, αυτού του κειμένου, αν δεν είχα αυτό το πρόβλημα υγείας θα το κάνω νωρίτερα. Αλλά το πρόβλημα υγείας σας σχετιζόταν με το φάκελο αυτό. Όχι, είναι μεγάλη, σοβαρή γρήπη. νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λείπει μία ψήφος. Έχει μείνει ένας που δεν ψηφίζει μια κάρτα μόνη της που έχει μπει αλλά δεν υπάρχει ψήφος. Καλώς. Εγκρίνεται. Μία αποχή μόνο. Μόνικα. Σήμερα που είστε καλά λοιπόν, μπορείτε να μας μιλήσετε για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Προϊόντων. Εκεί δεν ψηφίζουμε. Η κυρία Χόλμαερ, εδώ δεν υπάρχει συναισθηματική φόρτιση. Είναι θετικό το ε, πρόσημο του φακέλου. Θα είμαι σύντομη. Πρόκειται για την λήξη της ε, συμβάσεως μισθώσεως στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα κτίρια αυτά είχαν μισθωθεί το 2007 και προχωρούσαν σε περαιτέρω μισθώσεις. Πρόκειται για ένα κτίριο μάλλον ακατάλληλο με πολλούς χώρους που δεν χρησιμοποιούνται. Ε, είναι αναγκαίο να γίνουν και πολλές εργασίες επισκευών κλπ. Και γι' αυτό το λόγο ο οργανισμός ΕΚΑ ανεζήτησε άλλο κτίριο, βρήκε ένα κτίριο το οποίο μάλιστα είναι και καλύτερο αλλά και φθηνότερο κατά 500.000 ευρώ τον χρόνο και είναι και καλύτερο λειτουργικά. 18.000 τετραγωνικά μέτρα, 11.000 τετραγωνικά μέτρα για γραφεία, 6.000 για ε, ε, ε χώροι ε, συνεδριάσεων υπάρχουν επίσης εστιατόριο και αποθηκευτικοί χώροι καθώς και χώροι στάθμευσης. Το μίστομα είναι 5,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και θα χρειαστεί να αναλυφθούν βέβαια και τα δαπάνε για τις επισκευές. Όμως το κτίριο είναι ήδη σε καλύτερη κατάσταση από το παλαιό. Θα χρειαστεί λοιπόν ένα ποσό 5 εκατομμυρίων για να ε, διαρρυθμιστεί εκ νέου το κτίριο, να επισκευαστεί κτλ. Όποιος θέλει περισσότερες λεπτομέρειες ε, θα είναι σύντομα στη διάθεσή σα η φάκελη. Σας ευχαριστώ Μόνικα. Νομίζω ότι φτάνουν πια τα ακίνητα. Η κυρία Γκρέσλε για τον τριμερή διάλογο για την απλοποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού. η κυρία Γκρέσλε. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε να βρω το ε, σχετικό σημείωμα. Τέταρτη συνεδρία στην τριμερούς διαλόγου στο Στρασβούργο. Διήρκεσε τρεις ώρες. Λάβαμε νέες προτάσεις διατυπώσεων για άρθρα τα οποία είχαμε ήδη επεξεργαστεί καταλήξαμε σε μια προσωρινή ε, ρύθμιση για το 2, 6 και 7 για το blending, budget implementation και volunteering. Και μιλήσαμε για σχεδιασμένες και μη σχεδιασμένες μεταφορές πιστώσεων για οργανισμούς. Μιλήσαμε για έσοδα από χώρες ΕΖΕΣ Έχουμε το 34-2 για ε, άλλα σημεία του προϋπολογισμού, για την δημοσιονομική πειθαρχία που ήταν και μεγάλη ε, επιθυμία του Συμβουλίου και μετά από κάποιους σταθμούς τα δεχθήκαμε. Έχουμε το 39 3 α με νέο πίνακα για τα προβλεπόμενα των δαπανών των χωρών μελών και τα άρθρα 42, 3 και 4 για άλλα θέματα. Άρα, συζητήσαμε επίσης τα άρθρα 85 έως 89 και 91. Ολοκλώσαμε τη συζήτηση ορισμένων άρθρων για τις ευθύνες των οικονομικών φορέων. Και άλλο άρθρο που δεν είχε συμφωνηθεί στους αρχικούς τρεις τριμερείς διαλόγους, υπενθυμίζω άρθρο 2 με περιλαμβάνει ορισμένους ορισμούς και τον σημαντικό ορισμό του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, multiplier effect. το ερώτημα είναι εδώ αν θα καταφέρουμε να καταστήσουμε σαφείς τις ιδιωτικές επενδύσεις. Θα πρέπει εκεί να λάβουμε τον ορισμό του ΩΣΑ, διότι ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έως τώρα περιλαμβάνει μόνο τα δημόσια κονδύλια. Αν όμως δημόσια κονδύλια προσελκύουν άλλα δημόσια κονδύλια ή από δημόσιες τράπεζες, αυτό δεν μας ικανοποιεί για τα άρθρα 13 και 14 για τα decommitments, για το άρθρο 15 για τα προσωρινά δωδεκατημόρια σε περίπτωση μη συμφωνίας του προϋπολογισμού. Έχουμε επίσης το άρθρο 24 για το sponsoring, 37 για τις μεταφορές και την διατήρηση των εξουσιών του Κοινοβουλίου, 31 37 SMART Objectives και Impact Assessments και άλλα άρθρα όπως το άρθρο 36 για τις υποχρώσεις δημοσιεύσεως 49 αποθεματικό κρίσεως 54 διαβούλευση με τους πολίτες 57 service level agreements αποστολές σε ευρωπαϊκές πρεσβείες συγκρούσεις συμφερόντων με μελών κυβερνήσεων που διαχειρίζονται κοινοτικά χρήματα, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εθνικές δηλώσεις και συνδυασμό κονδυλίων από την περιφερειακή πολιτική. Άρθρο 62α1, ενιαίος κατάλογος ρυθμίσεων, παραμένει επίσης ανοιχτό εκεί, 63 ευρωπαϊκοί οργανισμοί, εκτελεστικοί οργανισμοί, 73 οι αρμόδιοι για, την, για τις υπογραφές και το τμήμα performance το οποίο αφορά πλήωνα άρθρα και συζητούμε αυτή τη στιγμή αν θα εξετάσουμε για τις δημοσιονομικές παρατυπίες και ε, πειθαρχικές διώξεις. Η επόμενη συνάντηση του τριμερούς διαλόγου θα γίνει την επόμενη Δευτέρα, όπου θα συζητηθούν και πάλι τα ανοιχτά θέματα για τα άρθρα που προανέφερα, καθώς και το κείμενο από το άρθρο 91 και μετά. Μέχρι τέλος του Νοεμβρίου προβλέπονται άλλες τρεις συναντήσεις τριμερούς διαλόγου και άλλες συναντήσεις μέχρι τέλους του έτους. Θα κάνουμε σχετική ανακοίνωση το συντομότερο δυνατό. Είναι σωστό λοιπόν να ανοίγονται οι φάκελοι αυτοί. Κάτι βέβαια ε, έχετε χάσει ως τώρα εσείς αλλά όχι πολλά. Προχωρούμε με το Συμβούλιο με την αναγκαία σοβαρότητα και θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και τις διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο με την ίδια αναγκαία σοβαρότητα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και η συγγήτρια. Ο κύριος Άσχορθ συμφωνεί μαζί σας. Ποιος επιθυμεί να παρέμβει. Νομίζω και οι οι συμφωνούν με την κυρία Γκρέσλε. Άλλος κανείς θέλει να βάλει το λόγο. Βλέπω ότι σας παθιάζει το θέμα. Ωστόσο, οι επιπτώσεις είναι σημαντικές. Θα πούμε στην κοινή γνώμη ότι έχουμε απλουστεύσει τον κανονισμό και θα δείτε την χαρά που θα ακτινοβολούν τα πρόσωπα όλων των πολιτών μας. Καλώς λοιπόν. Εν συμπεράσματι κυρία, κυρία Γκρέσλε. Ναι, συνεχίζουμε. Μιλούμε για 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν ε, είναι και μικρό ποσό. Αυτό είναι το πρόβλημα εν τέλει. Απλουστεύσεις ναι, αλλά υπέρ τίνος. Απλούστευση υπέρ των δικαιούχων, σύμφωνοι για τους ανθρώπους που χρειάζονται τα ευρωπαϊκά χρήματα για να δουλέψουν επί τόπου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε και το θέμα των εξειδικευμένων κανονισμών. Και τώρα συζητούμε τον κανονισμό Omnibus ελπίζω ότι θα μπορέσουν να γίνουν σημαντικά βήματα για την απλούστευση. Νομίζω ότι αυτά που μπορούμε να κάνουμε εδώ στο επίπεδο του θεσμικού μας οργάνου το κάνουμε ήδη. Αλλά εν τέλει είμαστε και υπόλογοι απέναντι στον φορολογούμενο. Μακάρι να μην είχαμε 725 τροπολογίε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, προσέξτε, το Συμβούλιο έχει καταθέσει 1200. Νομίζω λοιπόν ότι αξίζει τον κόπο η προσπάθεια και χαίρομαι πάντα όταν έχω κοντά μου και τους σκιώδεις συγητές. Θαυμάζω πάντως, λέει ο Πρόεδρος, τη δέσμευση των δυο ε, και ε, από τι οφόρο τιμής και στη γνώση και επιμονή ιδίω της κυρίας Κρέσλε. Καλά λοιπόν. Ε, έχοντας υπόψη και την χρονική στέρηση που μας κόστησε η ακρόαση του κυρίου ε, Βερχόφστατ, πάλι καλά που τελειώνουμε 12.30 και πριν από τις 12.30. Άψογα. Αρκούμεθα σε αυτά. Συνεχίζουμε στις 3. Θα προεδρεύσει ωστόσο ο κύριος Μουρεσάν, γιατί εγώ έχω να συμμετάσχω στις εργασίες της Επιτροπής Γεωργίας. Να με συμπαθάτε λοιπόν, αλλά θα επανέλθω μόλις τελειώσει αυτή η μου υποχρέωση. Διακόπτη τη συνεδρίαση.